εγκρίνεται. Προφορική τροπολογία έχουμε. Του κυρίου Μπουτικόφα. Έχετε το λόγο κύριε Μπουτικόφα. Κυρία Πρόεδρε, συνάδελφοι, θα ήθελα να κάνω την εξής πρόταση, προφορική τροπολογία, εκφράζει την πεποίθηση ότι η συμμετοχή της Ρωσίας στο Συμβούλιο της Ευρώπης είναι σημαντικό στοιχείο του παρόντος τοπίου θεσμικών σχέσεων στην Ευρώπη ελπίζει ότι πρέπει να βρεθεί τρόπος να πιστεί η Ρωσία να μην εγκαταλείψει ε, τη συμμετοχή της, να είναι μέλος του Συμβουλίου της Ευρώπης. Ευχαριστώ. Ψηφίζουμε την... Τι είπατε? Υπάρχουν αντιρρήσεις, συγγνώμη, υπάρχουν αντιρρήσεις ενστάσεις όσον αφορά την προφορική τροπολογία. Όχι. Ναι. Λοιπόν, ψηφίζουμε τώρα την προφορική τροπολογία υπέρ. Κατά αποχές, ας ελέγξουμε. Έλεγχος όσον αφορά την προφορική τροπολογία. Πέρας του έλεγχου. Εγκρίνεται. Οπότε πάμε στο ψήφισμα, στο σύνολό του, μέσω ονομαστικής ψηφοφορίας που ξεκινάει. Πέρας. Εγκρίνεται. Έχουμε έκθεση τη ΚΕΣΠΟΣΤ για τον άπτυξη ικανό τη Ευρωπαϊκή Ένωση για την πρόληψη συγκρούσεων και τη διαμεσολάβηση. Τροπολογία 1 υπέρ. Κατά. Αποχέ. Εγκρίνεται. Τροπολογία 2 υπέρ. Κατά. Αποχέ. Εγκρίνεται. Τροπολογία 3. Ονομαστική κλίση. Άρχεται. Πέρα. Εγκρίνεται. Τροπολογία 4. Ονομαστική κλίση. Άρχεται. Πέρας. Απορρίπτεται. Τροπολογία 5, ονομαστική κλίση, άρχεται. Πέρας. Απορρίπτεται το ψήφισμα στο σύνολό του με ονομαστική κλίση. Ξεκινάει. Πέρας. Εγκρίνεται λοιπόν. Ευχαριστώ συνάδελφοι. Εδώ ολοκληρώσαμε τον κατάξιο φοριών. Προχωρούμε σε ένα λεπτό στις επεξηγήσεις ψήφων. Colleagues, please, if you could leave the chamber, we could begin our... Παρακαλώ να αποχωρήσετε ήσυχα από την αίθουσα για να προχωρήσουμε στο επεξηγήσεις ψήφου. Πάμε λοιπόν στις επεξηγήσεις ψήφων. Θα ξεκινήσουμε με την έξηγη χάτουλα εθελοντική συμφωνητερική σχέση τη Ευρωπαϊκής Ενώσεως Βιετνάμ. Ο κύριος Κέλλη, έχετε το λόγο κύριε Κέλλη. Σα ευχαριστώ. Είναι καλό να είμαι πρώτο, κύριε Πρόεδρε. Καλωσορίζω αυτή τη σημαντική συμφωνία. Επενώ το έργο τη κυρία Χαουτάλα και του Φρανκ Πρόσ του συναδέλφου, η προστασία τη δασοκομεία και των δασών είναι σημαντικότατο στοιχείο όσον αφορά τη γενική προστασία του περιβάλλοντο και ε, μειώνει τη συνέπειε αλλαγή του κλίματο. Λοιπόν, θα πρέπει να αποφύγουμε την αποδάσωση και γι' αυτό καθορίζω αυτή τη σύσταση. Είναι ένα βήμα προ σωστή κατεύθυνση και για την Ευρωπαϊκή Ένωση και για το Βιετνάμ. Η διαφύλαξη των βιοτόπων και η βιοπικιλότητα μόνο μπορεί να επιτευχθούν μέσω τη συνεργασία με τρίτε χώρε για να εξασφαλίσουμε όχι μόνο ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν εξαγάγει παράνομη ξυλία, αλλά παρομοίω δεν υποστηρίζει το εμπόριο εισαγόμενου παράνομου υλικού ξυλία. Ελπίζω αυτή η θελοντική συμφωνία να πετύχει αυτό το στόχο και επίση τη δεσμεύση έλαβε το Βιετνάμ για να δημιουργήσει τι αναγκαίε δομέ για να συμπεριληφθεί να συμμορφωθεί με τη συμφωνία κάτι Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο κύριος Χάναν έχει το λόγο τώρα. Σας ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Είναι λογικότατη αυτή η συμφωνία για την Ευρωπαϊκή Ένωση, ούτω ώστε συνεργάζεται με το Βιετνάμ όσον αφορά τη βιωσιμότητα. Ρωτώ όμω τα μέλη, παρακαλώ τα μέλη να εξετάσουν το θαύμα που κατήστασε δυνατό τον να υπάρξει αυτή η έκθεση που εξάγει το αντίστοιχο του ΑΕΠ. Ε, το, το δεκαετία του 80 το Βιετνάμ ήταν από τις φτωχότερες ε, χώρες στον κόσμο. Λίγο πάνω από τα 200 δολάρια κατά κεφαλή. Τώρα έχει αυξηθεί το βιωτικό επίπεδο κατά 2.000% αν δούμε ποια είναι αγοραστική δύναμη και ισοτιμία ανάλογη. Εξαιρετική κατάσταση. Αν σκεφτούμε Πόσε προσπάθειε έκαναν οι ΗΠΑ για να εξαλείψουν με στρατιωτικού τρόπου τον κομμουνισμό. Ένα τρισεκατομμύριο δολάρια εξόδεψαν, 60.000 στρατιώτε χάσαν, 250.000 νοτιο χάθηκαν, ένα εκατομμύριο βορειοβιετναμίτε. Και απέτυχε ο πόλεμο. Και παρόλα αυτά, μετά από δύο δεκαετίε ελευθερίου, ελεύθερου εμπορίου, έχουμε φτάσει να επικρατεί το κράτο δικαίου και να υπάρξει ελεύθερο οικονομικό εμπόριο και οικονομία στη χώρα. Αυτό είναι το μάθημα. Α θα πρέπει να περνάνε τα αγαθά και υπηρεσίε στα σύνορα για να μην χρειάζεται να κινηθούν οι στρατιώτε. Πάμε στην επόμενη έκθεση Χάουτα, αλλά από αυτή τη φορά ασχολείται με το ψήφισμα για την Θελοντική Συμφωνία Ευρωπαϊκή ως Βιετνάμ. κυρία Μάγερ έχει το λόγο. Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Η Βρετανία είναι ο μεγαλύτερο αγωγέα τροπική ξυλία στην Ευρωπαϊκή Ένωση και σε σημαντικό βαθμό υποστηρίζω την εθελοντική αυτή συμφωνία με το Βιετνάμ. Είναι σημαντική συνεισφορά όσον αφορά την καταπολέμηση τη παράνομη ξυλία. Με την κυβέρνηση, η κοινωνία των πολιτών και τι επιχειρήσει να συνεργάζονται. Δυστυχώ, όλο τον κόσμο περίπου το μισό τη ξυλία προέρχεται από παράνομε πηγέ ε, το, το, η θελοντική προσέγγιση δεν θα νικήσει την παράνομη ξυλία, η Εγώ πιστεύω ότι το ΕΒ και η ΕΕ θα προχωρήσουν περισσότερο με νομοθεσία απαγορεύει την εισαγωγή παράνομη ή καταστρεφικά ε, αποκτημένη ξυλία. Θέλουμε μεγαλύτερη υποστήριξη, ούτω ώστε να εξαλειφθεί η διαφθορά όσον αφορά τι χώρε που παράγουν ξυλία. Η διαφθορα στον αφορα τι χωρε που λοτομία σε, και κοινότητε και κυβερνήσει χάνουν χρήμα, καταστρέφεται το οικοσύστημα, επιταχύνονται οι αλλαγέ του κλίματο και τελικά τροφοδοτούν συγκρούσει. Δεν θα πρέπει ε, να επαναπαυθούμε μέχρι η αγορά για παράνομη συλλία στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχει κλείσει για πάντα. Ευχαριστώ. Τώρα προχωράμε στην έκταση Dalton όσον αφορά ανταλλαγή πληροφοριών, όσον αφορά υπηκό των χωρών. Για ένα λεπτό, ο κύριο Τρογεύσκη έχει το λόγο. Ευχαριστώ. Η σημερινή συζήτηση ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρουσα και κατά τη διάρκεια τη συζήτηση ήμουν σε θέση να λάβω το λόγο σχετικά με το πρώτο τμήμα τη εκθέσεω. Δεν υπήρχε επαρκέ χρονικό διάστημα για να αναφερθώ στο δεύτερο θέμα, που είναι εξίσου σημαντικό και γι' αυτό θα ήθελα να συμπληρώσω τη χθεσινή μου παρέμβαση σήμερα. Το πιο επίμαχο θέμα ήταν η συμπερίληψη ε, ανθρώπων που έχουν διπλή υπηκότητα και με τα χαράς βλέπω ότι στο τέλος του 2019 καταφέραμε να καταλήξουμε σε κάποια συνεννόηση σχετικά με αυτό και οδηγηθήκαμε στη σημερινή ψηφοφορία. Επίσης θα ήθελα να πιστήσω την προσοχή σας και σε κάτι άλλο, σε ένα σημαντικό θέμα για εκείνους που δεν έχουν μόνο διπλή υπηκότητα, αλλά είναι και εκείνοι που μέχρι τώρα έχουν ε, αποφύγει τα προβλήματα που αφορούν το μητρό ε, σαν να απέφυγαν να μπουν στο Μητρό, και το Μητρό να μην ήταν σημαντικό για ποινικά θέματα. Εποφελή συμφωνία έκθεση Σοϊτρόβα για το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης και Σχετικό Πρόγραμμα. Η κυρία Μπίλντ έχει το λόγο. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Από την αρχή έλεγα ότι έχει βουλημικέ τάσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή που μαζί με το Ευρωπαϊκό Σώμα τη Αλληλεγγύη δημιουργεί επικάλυψη τη ε, θελοντική υπηρεσία. Δεν υπήρχε αμφιβολία ότι αυτό το νέο πρόγραμμα προσπαθούσε να δικαιολογήσει την ύπαρξή του επεκτηνόμενο συγνέχεια στον φάτα προνόμια του. Σήμερα όλα αυτά επιβεβαιώνονται. Λοιπόν, ενώ το προηγούμενο κείμενο υιοθετήθηκε μόλι πριν από μερικού μήνε, το πεδίο δράσεω επεκτάθηκε για τι επιχειρήσει ανθρωπιστική βοήθεια ε, όταν είναι ένα πολίτη ενό κράτου μέλου, δεν είναι πλέον προπόθεση να συμμετάσχει και αυξήθηκε ε, το προπολογισμό παράλογο. Όταν ξέρουμε το πρόγραμμα, δεν έχει την επιτυχία προβλεπόταν. Αυτό που μου, με απογοητεύει πολύ είναι η αδυναμία αυτέ οι δραστηριότητε τη αλληλεγγύη να γίνονται στη χώρα του καθενό. Οι Βρυξέλλε, λοιπόν, α, ήθελε να είναι αλληλέγγυα, αλλά όσο πιο μακριά από τον εαυτό τη μπορούσε. Και μα λέει ότι οι δραστηριότητε θα πρέπει να τονίζουν περισσότερο το ε, το προβλήμα που αντιμετωπίζουν μετανάστε. Το βλέπουμε. Είναι ένα ε, ένας κόσμος που κινείται για του άλλου. Ε, αρνούμενος κανεί τον εαυτό του. Αυτά. Ευχαριστώ. Ο κ. Μάμικιν. Ευχαριστώ πάρα πολύ κυρία Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι. Πιστεύω ότι το σώμα τη αλληλεγγύη έχει πραγματικέ δυνατότητε να δώσει ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία στι κοινωνικέ πολιτικέ. Ε, να δημιουργηθεί αλληλεγγύη μεταξύ τη Ευρωπαϊκή Νεολαία ε, και επιτρέπεται η προσωπική ανάπτυξη συμμετοχόντων. Είναι ιδιαίτερα υπέροχο ότι μετά το 2019 η οργάνωση από μη χώρε τη Ευρωπαϊκή Ενώση μπορεί να συμμετάσχουν σε αυτά τα προγράμματα σε περίπτωση τη πολιτική τη Ευρωπαϊκή Γειτονία. Αυτό είναι ένα άλλο στοιχείο στην αλυσίδα επαφών και επαφή και διπλωματία ανθρώπων με ανθρώπου. Πέραν αυτού, εδώ ενισχύουμε τη συμμετοχή των νέων και οι νέοι εκτιμούν ε, την άλλη πλευρά του έργου τους. Υποστήριξα αυτή την έκθεση και ε, μακάρι ο θελοντισμός να γινόταν ένα κομμάτι της ζωής και άλλων ομάδων πολιτών που θέλουν να συμμετάσχουν σε θέματα κοινοφελών συμφερόντων και να φροντίζουν τους άλλους, να μάθουν να φροντίζουν τους άλλους. Ευχαριστώ κύριε Ευχαριστώ. Θέλω να αναφερθώ σε τρία θέματα σήμερα. Πρώτον, οι προοπτικές ε, για το 2019 και 2020 αποτελούν απλώς έναν προσανατολισμό. Άρα θα πρέπει να ακολουθηθεί ο προσανατολισμός αυτός από έλεγχο. Επίσης, δεν ε, έχουμε εχέγγυα για την εύρυθμη λειτουργία των μελλοντικών προγραμμάτων. Επίσης, είναι πολύ σημαντική η χρήση νέων διάβλων επικοινωνία όπω τα κοινωνικά μέσα δικτύωσης. Είναι απαραίτητο όρος για την εφαρμογή αυτών των προγραμμάτων, γιατί διαφορετικά ε, δεν θα έχουμε την ε, επιδιωκόμενη επιτυχία. Μιλάμε για νέους ανθρώπους εδώ. Επομένως, πρέπει να υιοθετήσουμε νέες καινοτόμε στρατηγικές οι οποίες θα αντιστοιχούν στις συνήθειε και τις προτιμήσεις των νέων γενεών, ώστε το Σώμα αλληλεγγύη να μπορέσει να αποτελέσει πραγματικό τμήμα αυτών των προγραμμάτων για την συμβολή στην Ευρωπαϊκή Αλληλεγγύη. Ο κύριο Σάινφελ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύη δεν είναι απλώ μια εξαίρετη ιδέα είναι μια πραγματικά αξιόλογη πρωτοβουλία γιατί έχει εκπαιδευτικό χαρακτήρα, ηθικό χαρακτήρα, πλεονεκτήματα από άποψη ιδεοντολογίας και διαπαιδαγώγηση των πολιτών. Δεν μιλάμε λοιπόν απλώς για την προώθηση συγκεκριμένων ιδεών, αλλά για την υποστήριξη προς τους πολίτες να αναπτύξουν συγκεκριμένες δεξιότητες, να τους δοθεί η δυνατότητα ε, να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα ενεργά. 350.000 άνθρωποι θα συμμετάσχουν συνολικά στο πρόγραμμα. Στο το Ίδρυμα Καινοτομίας της Βιέννης ε, μάλιστα επένεσε αυτή την πρωτοβουλία και γι' αυτό και εγώ την υπερψήφισα. Κύριο Φαρία, ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Εγώ υπερψήφισα την ε, έκθεση αυτή για την ε, δημιουργία του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης. Σε καιρούς λαϊκισμού και εθνικισμού εγώ ε, υποστηρίζω οτιδήποτε ε, ενισχύει την αλληλεγγύη και την συνεργασία των πολιτών. Ε, είναι πραγματικά ε, μια εξαιρετική ευκαιρία που δίνεται μέσα από το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης να αποκτήσει κανείς νέες επαγγελματικές δεξιότητες σε πολύ σημαντικούς Τομεί, Είναι πάρα πολύ σημαντικό η υλοποίηση αυτού του προγράμματος να μην συνοδευτεί από καταχρήσει απλώς για να ε, εκμεταλλευτούν μη κυβερνητικέ οργανώσεις ή και κρατικοί φορεί φθηνό εργατικό δυναμικό. Πρέπει όσοι συμμετέχουν να έχουν ε, ε, δίκαιη και επαρκή αμοιβή για αυτά που θα κάνουν. Ευχαριστώ, κύριο Σκέλη. Σας ευχαριστώ και εγώ υπερψήφισα την έκθεση αυτή. Η στόχοι αυτού του προγράμματος, του σημαντικού αυτού προγράμματος για την προώθηση της αλληλεγγύης μεταξύ των πολιτών και τη συμμετοχή των νέων. Το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης είναι ένα εξαιρετικό δρόμος ώστε οι νέοι να αναπτύξουν τις ε, δεξιότητες τους μέσω από πρακτικέ ασκήσει, μαθητείε για την απόκτηση πραγματικών εμπειριών. Το πρόγραμμα αυτό και η επέκτασή του θα δώσει τη δυνατότητα σε πολλού περισσότερους νέους να το εκμεταλλευτούν, να το αξιοποιήσουν και θα βοηθήσει στην ένταξη περιθωριοποιημένων ε, νέων. Ήδη ε, εκατοντάδες Ιρλανδοί νέοι έχουν ε, δηλώσει τη συμμετοχή τους. Ελπίζω να αυξηθούν, ιδίως στις ε, περιοχές της Υπέθρου και σε άλλες μειονεκτούς περιοχές που επίσης είναι ιδιαίτερος στόχος των, του προγράμματος αυτού. Σας ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Ευχαριστώ. Περνάμε στην έκθεση Νίμπλερ για την κυβερνοασφάλεια. Ο κύριος Μαριάς. Μιλούμε για την κυβερνοασφάλεια τη στιγμή που υπάρχουν σοβαρές παραβιάσεις σε συγκεκριμένα κράτη μέλη. χθες ζήτησα από τον επίτροπο τον κύριο Άνσιπ, να τοποθετηθεί στις καταγγελίες που έκανα διότι η ελληνική κυβέρνηση προβαίνει σε προληπτικές συλλήψεις όσων διαφωνούν με το ξεπούλημα της μακεδονίας μας και της ιστορίας μας και έκανε προληπτικές συλλήψεις στην περιοχή των γιαννιτσών. είπε δε η υπουργός προστασίας του πολίτη ότι γνωρίζει τα στοιχεία τους διότι παρακολουθεί η αστυνομία το facebook και τα social media. αυτό συμβαίνει σήμερα στην ελλάδα και σχηματίζονται δικογραφίες εναντίον όσων διαφωνούν με το ξεπούλημα της μακεδονίας όσων διαφωνούν με την κατάπτυστη συμφωνία των πρεσπών όσοι συμμετέχουν στα συλλαλητήρια και η κυβέρνηση επεξεργάζεται τα προσωπικά της δεδομένα και παρεμβαίνει και βλέπει τι υποστηρίζουν και τι λένε στα social media. πρέπει να υπάρξει τοποθέτηση της κομισιόν για το θέμα αυτό. Κύριε Στρογεύσκη. Ευχαριστώ. Είναι πολύ σημαντικό το θέμα αυτό και πρέπει να μην χάσουμε χρόνο. Ε, οι διαδικασίε ξεκίνησαν πριν από δύο χρόνια. Να σα υπενθυμίσω ότι τον Δεκέμβριο πέρσι επιτέθηκε συμφωνία στο πλαίσιο του τριμερού διαλόγου και το αποτέλεσμα αυτού ήταν τον Ιανουάριο η Επιτροπή Ήτρε να επιβεβαιώσει ε, την ε, κατεύθυνση που είχε χαρακτηρίσει και σήμερα ψηφοφορήσαμε. Η μόνιμη εντολή του οργανισμού έχει πολλά πλεονεκτήματα Εκτός από τη συλλογή πληροφοριών και δεδομένων και την εμπειρογνωμοσύνη, για πρώτη φορά έχουμε τη δυνατότητα να προχωρήσουμε σε επιχειρησιακές δραστηριότητες. Και θέλω να πιστήσω την προσοχή σας σε αυτό το γεγονός, διότι η κυβερνοασφάλεια είναι ένας τομέας όπου πραγματικά είναι πάρα πολύ σημαντικό να αναλαμβάνεται δράση και όχι μόνο να συλλέγονται δεδομένα. Πρέπει η δράση να είναι εκείνη που εξασφαλίζεται κατά προτεραιότητα. Ο κύριο Κέλλη. Ε, σας ευχαριστώ. Εγώ υπερψήφισα την ε, έκθεση αυτή. Συμμετείχα και χθε στη σχετική συζήτηση που προηγήθηκε και θέλω να συγχαρώ για άλλη μια φορά την φίλη και συνάδελφο Αγγέλικα Νίμπλερ για το εξαιρετικό της έργο. Κάθε μέρα ακούμε στις ειδήσει για κυβερνοεπιθέσεις που γίνονται είτε από μεμονωμένα άτομα είτε και από εγκληματικές οργανώσεις. που πολλές φορές προέρχονται και από χώρες όπως η Ρωσία ή η Βόρεια Κορέα. Πρέπει λοιπόν να υπάρχει επαγρύπνηση για να καταπολεμηθούν τέτοιου είδους επιθέσεις. Ιδιαίτερος χαιρετίζω τις ε, αρμοδιότητες που ανατίθενται στον ΕΝΙΣΑ και τις δράσεις που θα μπορεί να αναλάβει ο οργανισμός στη βάση της ε, πράξης που συζητήσαμε. Θεωρώ ότι είναι ένα, ένα βήμα στη, στη σωστή κατεύθυνση. Έκθεση ε, ε, Κάστρο για τις αθέμενες πρακτικές στην αλυσίδα τροφίμων. Μιράντα. Ευχαριστώ πολύ. Υπερψήφισα την έκθεση αυτή, γιατί γνωρίζουμε ότι η χώρα μου όπου κάνει 80 σαντίμ το λίτρο το γάλα, δεν ε, κερδίζουν ε, οι παραγωγοί παρά το κόστος παραγωγής τίποτα παραπάνω. Είναι λοιπόν σε κατάσταση αδυναμίας με αθέμητες εμπορικές πρακτικές. Δεν καταφέρνουν να διαπραγματευτούν όπως θα έπρεπε ώστε να αγοράζουν σωστά τα προϊόντα τους ε, οι καταναλωτές. Και η Ευρωπαϊκή Ένωση τελικά θα έπρεπε να παρέμβει και το έκανε τρεις φορές μέχρι τώρα εξαιτίας ακριβώς της κατάστασης. Και τώρα λοιπόν και πάλι. Γι' αυτό και η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τις αθέμητες εμπορικές πρακτικές προκειμένου να στηρίξουμε τον γεωργικό πληθυσμό. Ξέρουμε ότι οι αγρότες χρειάζονται περισσότερη προστασία από αυτές τις αθέμητες εμπορικές πρακτικές. Ευχαριστώ. Κύριος Μαριάς. Προκειμένου να στηριχθούν οι αγρότες μας πρέπει να υπάρξει απόλυτη απαγόρευση όλων των αθέμητων πρακτικών και όχι μόνο συγκεκριμένες πρακτικές όπως περιγράφει η έκθεση. Όλες οι πρακτικές που είναι αθέμητες πρέπει να σταματήσουν διότι είναι δεδομένο ότι οι παραγωγοί κερδίζουν μόνο το 20% επί της τιμής πώλησης ενός αγροτικού προϊόντος διότι επί της ουσίας υπάρχει αισχροκέρδεια από την πλευρά των εταιριών διανομής τροφίμων από τις αλυσίδες διατροφής οι οποίες επί του πρακτέου εκμεταλλεύονται τους ίδιους τους παραγωγούς με εκβιασμούς με μείωση των τιμών παίρνουν επιταγές και στο τέλος δεν πληρώνουν και επίσης οι χονδρέμποροι επί της ουσίας διαμορφώνουν τέτοιες τιμές που οι ίδιοι οι παραγωγοί δεν έχουν κανένα κέρδος. άρα απόλυτη απαγόρευση όλων των αθέμητων πρακτικών που είναι εις βάρος των γεωργών μας. Ο Ευχαριστώ πολύ. όταν πληρώνεται κανείς 30 μέρες μετά, όταν ακυρώνονται παραγγελίες, όταν αλλάζουν οι όροι, οι καθυστερήσεις, όλες αυτές οι διαδικασίες έχουν σαν αποτέλεσμα τελικά να χαλάνε τα προϊόντα. Όλες αυτές οι πρακτικές αποτελούν παράδειγμα μόνο αθέμητων εμπορικών πρακτικών και είναι πολύ καλό που σήμερα ασχολούμαστε με αυτές. Και είναι επίσης καλό που πρόκειται για οδηγία και όχι για κανονισμό, γιατί έτσι οι χώρες μέλη έχουν ευελιξία προκειμένου να αποφασίσουν τι θα κάνουν. Πάντα βέβαια υπάρχουν δύο πλευρές σε μια σύμβαση και αν η μία πλευρά ασκεί αθέμητες πρακτικές απέναντι στο πιο αδύναμο, τότε κάτι θα πρέπει να γίνει για να επανέλθει δικαιοσύνη. Ευχαριστούμε. Περνάμε στην έκθεση Σέφλιν, Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών. Η κυρία Σκοτ Κέτο ήταν η πρώτη, δεν είναι εδώ όμως. Η κυρία Μιράντα έχει το λόγο. Παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε. Είμαι υπέρ της έκθεσης Σέπφλιν γιατί πιστεύω ότι η πρωτοβουλία αυτή η Ευρωπαϊκή Πολιτών αποτελεί ένα άμεσο εργαλείο για να ακούμε τους πολίτες οι οποίοι έτσι συμμετέχουν στη δημοκρατική διαδικασία. Υπήρξε η πρωτοβουλία για το δικαίωμα στο είδωρ που είναι βασικό αγαθό για τις ε, γλώσσες των μειονοτήτων και τα δικαιώματα των ανθρώπων που μιλούν τέτοιες γλώσσες. Πολλά μπορούμε ακόμα να κάνουμε για να συγκεντρώσουμε ε, υπογραφές και εκστρατείες για την ευαισθητοποίηση του κόσμου. Μέχρι τώρα λίγες πρωτοβουλίες εγκρίθηκαν όμως από τότε που ξεκίνησε η διαδικασία αυτή. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να προσφέρει ένα μητρό online στους πολίτες έτσι ώστε να μπορούν να διαχειρίζονται την πρωτοβουλία από την αρχή μέχρι το τέλος. Με ένα δημόσιο χώρο στο διαδίκτυο με γενικές πληροφορίες ε, συγκεκριμένε ε, όμως για το στόχο μας. Ευχαριστώ κύριος Μαριάς. Η Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών είναι μία έκφραση της αρχής της συμμετοχικής δημοκρατίας στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και θα πρέπει να ασκείται με τον πιο δημοκρατικό πιο άμεσο και ακόλιτο τρόπο χωρίς γραφειοκρατίες. εδώ υπάρχει μια αντίφαση. με την ευρωπαϊκή πρωτοβουλία οι πολίτες καλούν την κομισιόν να αναλάβει νομοθετική πρωτοβουλία. ποιος όμως είναι αυτός που ελέγχει αν η νομοθετική πρωτοβουλία αυτή των πολιτών είναι σύνομη; η κομισιόν. δηλαδή εδώ έχουμε γιάννη σπίνη και γιάννη σκερνάη δηλαδή πρακτικά τι συμβαίνει η ίδια η κομισιόν ελέγχει αν η νομοθετική πρωτοβουλία είναι ορθή ενώ η ίδια η πρωτοβουλία καλεί την κομισιόν να αποφασίσει. είχα πει ότι άλλο όργανο έπρεπε να ελέγχει την νομιμότητα της πρωτοβουλίας των πολιτών. σε κάθε περίπτωση χρειάζεται ένα σύστημα που να δίνει την ευκαιρία στους πολίτες ακόλυτα να ασκούν αυτό το δικό τους δικαίωμα το οποίο είναι δικαίωμα συμμετοχικής δημοκρατίας. ευχαριστώ. Ο κύριος Μάμεκινς. Ευχαριστώ, συνάδελφοι. Η Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών δημιουργήθηκε ως ένα εργαλείο για να δώσουμε περισσότερη εξουσία και συμμετοχή στους πολίτες στην ομοθετική διαδικασία. Δεν φτάνει όμως γιατί καμία νομοθετική πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής δεν βασίστηκε σε αυτή την πρωτοβουλία. 63% των πολιτών είτε δεν γνωρίζουν καθόλου, είτε ελάχιστα γνωρίζουν ποια είναι τα δικαιώματά τους βάσει της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας. Από την άλλη μεριά, διάφορα λόμπι δρούν στις Βρυξέλλες. Και αυτή είναι μια πραγματικότητα που έχει σαν αποτέλεσμα να δυσκολεύονται οι πολίτες να κάνουν τη φωνή τους να ακουστεί. Κατά τη γνώμη μου, το πακέτο μεταρρυθμίσεων δυσκολεύει ακόμα περισσότερο τους πολίτες να συμμετέχουν, γιατί ας πούμε περιορίζεται το σύστημα online για την συλλογή υπογραφών. Είμαστε όμως στον 21ο αιώνα και πρέπει ηλεκτρονικά να μπορούμε πολύ πιο εύκολα να λειτουργούμε. Γενικό όμως είμαι υπέρ και υπερψήφισα. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε κύριο Σένφελτ. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Κύριε Πρόεδρε, αυτή η Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών δεν αποτελεί μόνο ένα δημοκρατικό εργαλείο, αποτελεί και έναν ε, μηχανισμό ο οποίος επιτρέπει στους πολίτες να ενώνονται γύρω από μία ιδέα, γύρω από ένα θέμα, γύρω από ένα κοινό στόχο και σκοπό. Και νομίζω ότι αυτό που χρειάζεται είναι τουλάχιστον 7 πολίτες από 7 χώρες είναι η ελάχιστη περίπτωση και φυσικά χρειάζεται εκατομμύρια εκατομμύριο υπογραφές στη συνέχεια. Ε, χρειάζεται επίση περισσότερη ελευθέρωση για να γίνονται πιο εύκολα τα πράγματα σε αυτή τη διαδικασία. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, αποφάσισε να στηρίξει περισσότερο την πρωτοβουλία τη συλλογή υπογραφών ε, και να κάνει και άλλε βελτιώσει. Είναι σημαντικό πάντω το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να διαβουλεύεται. Είμαι υπέρ. Ευχαριστούμε. Ο κύριο Φαρία. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Είμαι υπέρ της έκθεσης αυτής. Είναι μια ευρωπαϊκή πρωτοβουλία που είναι απαραίτητη για να έρθουν πιο κοντά οι πολίτες στην Ευρώπη. Θα πρέπει να ενώσουμε περισσότερο τους πολίτες, όχι να τους διχάσουμε. Χρειαζόμαστε μια Ευρώπη που σίγουρα έχει διαφορές, αλλά πρέπει να διαθέτει και πλατφόρμες για συλλογή υπογραφών και από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αλλά και από ανεξάρτητους πολίτες. Σίγουρα χρειάζεται έλεγχος για να αποφεύγονται απάτες. Πρέπει όμως μια τέτοια πρωτοβουλία όπως αυτή να ενώνει την κοινωνία και να συμπεριλαμβάνονται εκεί όλοι οι παραγόντες της κοινωνίας και να αφήνουμε αρκετό χρόνο ώστε οι πρωτοβουλίες αυτές να προχωρούν και να καταλήγουν ε, σε νομοθετικές πρωτοβουλίες. Οι πολίτες θα πρέπει όπου και αν βρίσκονται στην Ευρώπη να μπορούν να συμμετέχουν. Δεν θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη τα συμφέροντα μόνο μιας χώρας ή μόνο ενός τμήματος ε, οικονομικών συμφερόντων. Πρέπει να χρησιμοποιείται σωστά το δημοκρατικό αυτό εργαλείο στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Η επόμενη έκθεση είναι η έκθεση της κυρίας Κανιέτε. Το λόγο έχει ο κύριος Μάμακενς. Αγαπητοί συνάδελφοι, εντυπωσιάζομαι από το εχθρικό πνεύμα με το οποίο έπνευσε αυτή την έκθεση ο συγγητής. Λέω ότι οι σχέσει Ευρωπαϊκή Ενώσεω και τη Ρωσία στην αποτροπή και την απομόνωση εδράζονται. Δίνει πολλέ συστάσει σχετικά με τον περιορισμό της συνεργασίας με τη Ρωσία και καμία σύσταση για την επανάληψη της επικοινωνίας. Επίσης υπονομεύει την αξιοπιστία του μηνύματος του Συνόσου εκφράζοντας απλώς πεπιθήσεις και καταδίκες για θέματα τα οποία δεν έχουν καν εξηχνιαστεί όσον αφορά τις κυρώσεις. Όσο πιο αποτελεσματικέ είναι για την αποδυνάμωση τη ρωσική οικονομία, τόσο ε, μειώνεται και επίτευξη του στόχου τη Ευρωπαϊκή Ενώση δεν είναι καλύτερο εταίρο έτσι η Ρωσία και οι κυρώσει περιθωριοποιούν και τα μέλη τη ρωσική ελίτ. Δηλαδή, χάνουμε συνομιλητέ που χρειαζόμαστε. Και βέβαια, πραγματική πρόξη Ευρωπαϊκή Ενώσεω όσον αφορά την εξωτερική πολιτική ε, δεν είναι τόσο η Ρωσία. Ελπίζουν με αντιπαράθεση κατά της Ρωσίας οι πολιτικοί να συλλέξουν κάποιες ε, ψήφους από εκεί κατά της Ρωσίας. Ο κύριος Νέκοφ. Ευχαριστώ, συνάδελφοι. Συμφωνώ με αυτά που είπε ο κύριος Μάμικινς. Η Ρωσία είναι μια χώρα στρατηγικής σημασίας για το μεγαλύτερο τμήμα της Ρωσίας. Έχει σύνορα με τα περισσότερα κατημέλη της Ευρωπαϊκή έχει ενό σύνορο με την Ένωση, με μήκος πάνω από 2.300 χιλιόμετρα. Είναι στρατηγικός ε, εταίρος και νομίζω ότι κάνουμε στρατηγικό σφάλμα διότι απορρίπτουμε την ε, ε, ρεαλιστική πολιτική του 21ου αιώνα. Δεν χρειάζονται πολιτικές διακηρύξεις ε, και πατοναλιστικός τόνος. Στην παράγραφο 26 καταδικάζεται η συμμετοχή της Ρωσίας στην, περίπτωση, στην υπόθεση Σκρυπάλ. Οι επίσημες υπηρεσίες του Ηνωμένου Βασιλείου δεν είναι ε, σίγουροι όσον αφορά τα συμπεράσματά τους και οι συνάδελφοι που στήριξαν το κείμενο αν έχουν περισσότερες πληροφορίες αυτοί από την Intelligence Service δεν ξέρω. επικρίνουμε τον ερευνητή, την ερευνητική δημοσιογραφία σε τρίτες χώρες, στη Βουλγαρία όμως απαγορεύονται εκπομπές λόγω των πληροφοριών που παρέχουν. Τελευταία έκθεση είναι η έκθεση για και δίνω το λόγο στην κυρία Μάγερ. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Οι ένοπλε σειράξει. πολύ σπάνια γίνονται ε, στο πεδίο τη μάχη, αλλά στι κοινότητε, η παιδεία, η υγεία, η απασχόληση, οι μεταφορέ όλοι υποφέρουν. Οι γυναίκε είναι το μέσο όλων αυτών, αλλά αποκλείονται στο έργο αποφυγή τη σύραξη και στη, να συμμετέχουν στη Μεσολάδευση διαμεσολάβηση και στην ίνευση. Είναι 2% των διαμεσολαβητών και 5% των μαρτύρων σε ειρηνευτικές διαδικασίες ή υπογραφών των μελών. Αυτή η έκθεση, όπως το ψήφισμα 1325 του ΟΗΕ, σωστά δέχεται ότι διαφορετική εμπειρία των γυναικών που σειράξει από ότι άντρε, όπω το Κασμίρ. 8.000 άντρε έχουν χαθεί, είναι αγνοούμενοι από το 2013 και μισέ χείρε ζουν στη φτώχεια, δεν έχουν δικαίωμα ιδιοκτησία και δεν μπορούν να ξαναπαντρευτούν αεροβόλα που τραυματίζουν και κροτηριάζουν και χρησιμοποιείται και ε, ο βιασμό σαν ένα όπλο πολέμου. Χρειάζεται τώρα νέα προσέγγιση και ελπίζω ότι αυτή η έκθεση είναι ένα βήμα προ τη σωστή κατεύθυνση. Ευχαριστώ κυρία μου. Εδώ ολοκληρώθηκε η επεξήγηση ψήφων. Διακόπτεται η συνεδρίαση μέχρι τις 3. Καλή σας όρεξη.